μπορέσετε να εκφράσετε τη γνώμη σας και να πείτε ότι ορίστε πραγματικά η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου ενδιαφέρθηκε, με ρήμνησε για αυτό το θέμα με θετικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Υφυπουργέ, λέει ο Πρόεδρος και έτσι μπορώ να, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε απόλυτη, απόλυτα πλήρη εμπιστοσύνη στην Ουγγρική Προεδρία και ε, μπορώ να πω ότι ολοκληρώνουμε εδώ τις συζητήσεις μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και η επόμενη συνεδρίασή μας θα διεξαχθεί αύριο που είναι πέμπτη ημέρα πέμπτη στις 9 το πρωί και το απόγευμα στις 15.00 στις 3 το απόγευμα έχετε ενημερωθεί σε σχέση με την ημερήσια διάταξη μπορείτε να την βρείτε και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας ευχαριστώ, γεια σας